Ο πρόεδρος έλαβε από την ομάδα ECR ένα αίτημα διορισμού σε επιτροπές και αντιπροσωπείες θα συμπεριληφθούν αυτά στα σημερινά συνοπτικά πρακτικά. Εάν δεν έχετε παρατηρήσεις μέχρι την έγκρισή τους, οι διορισμοί αυτοί θα ε, θεωρηθούν εγκεκριμένοι.